ένα διασυνοριακό σώμα που εκπροσωπεί διάφορες χριστιανικές ομολογίες στην ίσο της Ιρλανδίας, βορρά και νότο, ε, που βρίσκονται στο θεωρείο των επισήμων. Σα Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή και συμπίπτει να προεδρεύω. Ε, χαίρομαι. Θα ήθελα να προσθέσω ότι έχουν στι Βρυξέλλε επισκέπτε μα για να συζητήσουν με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα διάλογο που προβλέπεται από τις συνθήκες. Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι εκκλησίες στην Ίσο έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ευτική διαδικασία, κάτι που υποστήριξε στεναρά το Κοινοβούλιο μας. Μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε φιλοξενήσει μια πολύ θετική έκθεση ε, σχετικά με την ενευτική πρωτοβουλία και τη χρηματοδότηση της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλώς ορίσατε ε, και είναι πολύ επίκαιρη η επίσκεψή σας. Παρακαλώ να διαβιβάσετε στις κοινότητές σας ότι είναι πάγια υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Σόριν Μόισα εγκατέλειψε την ομάδα S&D, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, από τις 22 ε, Νοεμβρίου και ε, από τις 29 του μηνός σήμερα ανήκει στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η Επιτροπή